Η Οι αρχές της Λουθουανίας ε, μου απέφθηναν ένα αίτημα για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Βίκτορ Ουσπατσίκ στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαδικασίας ε, στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βίλνιου. Σύμφωνα με το άρθρο 6, Παράγραφό 2 του κανονισμού, το αίτημα αυτό το διαβίβασα στην Νομική Επιτροπή που είναι αρμόδια για το θέμα. Επίσης έλαβα από τις ομάδες ΕΛΚ πολλά αιτήματα τροποποίηση στι ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και τι διακοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείε. Ο κατάλογο αυτών των ε, ονομάτων θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Συνόδου. Εάν ε,